Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί Επιτροπή, να ξαναρχίσουμε την ε, συζήτησή μας. Θα ήθελα παρακαλώ όλοι να καθίσετε και ήσυχα. Θα περάσουμε τώρα σε μια επόμενη φάση μετά από αυτήν την γενική παρουσίαση των του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου βάσει των εισηγήσεων των κυρίων Ρεν και Άντορ θα περάσουμε τώρα στην εξέταση τριών θεμάτων. Το πρώτο σήμερα το πρωί θα αφορά τον κοινοτικό προϋπολογισμό και το συσχετισμό του με τους εθνικούς. Το έπειτα το θέμα των, του συντονισμού των εθνικών οικονομικών πολιτικών αυτό το μεσημέρι και μετά και έπειτα τις πολιτικές απασχόλησης. Να καλωσορίσω εδώ και εκπροσώπους της Κυπριακής Προεδρίας, λέει ο Πρόεδρος, και ο κύριος Λίντς θα πάρει το λόγο μετά τον Επίτροπο. Επίσης, χαιρετώ τον κύριο Λεβαντόφσκι, Επίτροπο Επιτροπολογισμού, που θα μας παρουσιάσει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κοινοτικό δημοσιονομικό πλαίσιο των επόμενων ετών. Παρακαλώ ησυχία. Και να θυμίσω ότι θα ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία. Όσοι θέλουν το λόγο να γράψουν το όνομά τους στον πορτοκαλί κατάλογο που μοιράστηκε Δεν λευκό είναι το χαρτί, να βάλουν το όνομά του το κοινοβούλιο από το οποίο έρχονται και τις αρμοδιότητές τους. ώστε να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε το χρόνο μεταξύ των χωρών και των πολιτικών ομάδων και των διαφόρων κοινοβουλίων. Κάποια λόγια είναι ήδη εισαγωγής τώρα για να σας παρουσιάσω τον ε, προβληματισμό που θα μας απασχολήσει κυρίως σε αυτή τη συζήτηση της Τρογγυλής Τράπεζας, αυτή τη συνάντηση. Θέλουμε να δούμε το συσχετισμό μεταξύ των ε, εθνικών και του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερο σημαντικό σε αυτή τη χρονική συγκυρία. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί όλοι οι εθνικοί μας προϋπολογισμοί περνάνε από μια προσπάθεια λιτότητας και επανεξισορρόπησης, κάτι που σε πολλές χώρες δεν έχει γνωρίσει κάτι τέτοιο στο παρελθόν ποτέ. 20 από τις 27 χώρες υπόκεινται σε διαδικασία για υπερβολικό έλλειμμα. 25 κράτη-μέλη στα 27 επίσης έχουν υπογράψει το σύμφωνο για την δημοσιονομική εξυγίανση που τέθηκε σε ισχύ στις αρχές του τρέχοντος μήνα. Επίσης, ακριβώς την ίδια στιγμή έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το ευρωπαϊκό, τον Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Προπολογισμό δηλαδή για την ερχόμενη επταετία και ελπίζουμε σύντομα μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα να καταλήξουμε σε συμφωνία βάσει των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, ο κοινοτικός προπολογισμό, θα αποτελέσει τον 28 ο θα αποτελέσει τον 28ο κοινοτικό προπολογισμό. 21 όταν προσχωρήσει και η Κροατία. Ένα μεγάλο μέρο ε, του κοινοτικού προπολογισμού προέρχεται από τι εθνικέ συνεισφορέ, του δικού σα προπολογισμού. Όμω το 94% των δαπανών του κοινοτικού προπολογισμού επιστρέφουν, επιστρέφουν στα κράτη-μέλη και έρχονται να ανακουφίσουν, να ενισχύσουν δηλαδή τους εθνικούς προπολογισμούς όπως με την πολιτική συνεργασίας με τις τρίτες χώρες και έτσι ο κοινοτικό προπολογισμό γίνεται ένας επιπλέον, ένας συμπληρωματικός προπολογισμό για τον καθέναν από τους εθνικούς από την πλευρά των εσόδων όσο και από την πλευρά των δαπανών. Η κρίση που διανύουμε εδώ και μια τριετία είναι ένας παράγοντας που έχει αποκαλύψει κάποια νέα στοιχεία. Και από τη μια πλευρά και από την άλλη δηλαδή. Έχει δείξει από τη μία πλευρά ότι υπάρχουν κοινά συμφέροντα μεταξύ των κορών και αυτό ήταν πολύ πιο ισχυρό στοιχείο από ό,τι φανταζόμασταν. Η αγαπητή μας Ιρλανδία εκπροσωπεί λιγότερο από το 1% των ε, κατοίκων, των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των καλύτερων ίσως, αλλά είναι 1%. Η Ελλάδα με ΑΕΠ που είναι το 2% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλα αυτά τα στοιχεία, η θέση των δύο, αυτό, ε, των δύο αυτών εταίρων μας απασχόλησε επί μήνες και δεν πρέπει να αποτίσω φόρο τιμής και στην Ιρλανδία και στην Ελλάδα που έκαναν τιτάνιες προσπάθειες για να ξεφύγουν από τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν. Η Ομοσπονδία της Γερμανίας πριν από δύο χρόνια αποφάσισε εξέφνης να πάψει τη χρήση, την παραγωγή μάλλον πυρηνικής ενέργειας στη χώρα. Αυτό είχε συνέπειες σε όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπηρέασε τις τιμές ενέργειας και την κατάσταση της ενέργειας. Πριν το τέλος του μήνα θα διεξαχθούν εκλογές στην Ιταλία. Δίνω κάποια παραδείγματα τυχαία και παράξενα. Ε, το πρόγραμμα που θα θέσει σε εφαρμογή η κυβέρνηση που θα εκλέγει από του Ιταλού πολίτε θα επηρεάσει την, την ζωή και την πολιτική όλων των εταίρων τη Ιταλία. Μιλάμε λοιπόν για μια κοινότητα συμφερόντων που έχει γίνει ένα κοινό πεπρωμένο. Ό,τι συμβαίνει στη χώρα του ενό έχει θετικέ ή αρνητικέ συνέπειε για τι υπόλοιπε χώρε. Και από την άλλη πλευρά, η κρίση μα έδειξε επιπλέον ότι δεν διαθέτουμε μηχανισμού αλληλεγγύη ή στο ύψος ακριβώς ε, των απαιτήσεων αυτών των κοινών συμφερόντων. Βεβαίως έχουμε προβλέψει κάποια ταμεία όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Αλληλεγγύης αλλά για να κάνω και μια σύγκριση με το χώρο της υγείας είναι σαν ένα σαν μηχανικό αναπνευστικό μηχάνημα. Δεν πρόκειται για μια οριστική θεραπεία. Κάποιοι από εσά σήμερα το πρωί, εκπρόσωποι από την Ισπανία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Κύπρο και την Λετωνία, επιμείνατε στο γεγονός ότι πέραν της δημοσιονομικής πειθαρχία που απαιτείται, πέρα από την βοήθεια που θα προσφέρει ο μηχανισμός αλληλεγγύης και άλλου τέτοιου είδους ε, συστήματα, θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε τις ε, επενδύσεις για το μέλλον, απαραίτητες για την ε, επιστροφή της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας. Χωρίς την ανάπτυξη δεν θα υπάρξει λύση ούτε στο πρόβλημα του χρέους, ούτε των ελλημάτων, ούτε της ανεργίας. Έτσι, εφόσον στις 28 δημοσιονομικές μας πολιτικές οφείλουμε να συνδυάσουμε τους περιορισμούς, τη μείωση των ε, διοικητικών δαπανών που απαιτούνται και ταυτόχρονα να διατηρήσουμε τις επενδύσεις για το μέλλον, τις απαραίτητες δαπάνες για το μέλλον, θα πρέπει από κοινού να θέσουμε κάποιες ερωτήσεις για να προσπαθήσουμε να βρούμε απαντήσεις για το τι προσδοκούμε όλοι από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό τι περιμένουμε από την πλευρά των δαπανών, πώς θα μπορούσαν να ενισχύσουν, να συμπληρώσουν τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Υπάρχουν πολιτικές κατάλληλες ώστε η κρίσιμη μάζα των δαπανών να οριστεί και να πετύχουμε την οικονομική αποτελεσματικότητα που αναζητούμε, την ευρωπαϊκή προστεθέμενη αξία, όπως μας είπε και ο εκπρόσωπος της Βουλής των Λόρδων σήμερα το πρωί. Είναι λογικό να αφιερώνουμε στον ευρωπαϊκό προπολογισμό πενταπλάσια κονδύλια για τη γεωργία από ό,τι για το μέλλον της ανάπτυξης και της έρευνας. Τέθηκαν ερωτήσεις το πρωί για την αρχή της επικουρικότητας από τον κύριο Βαντερλίντεν, για παράδειγμα, ή για την περιφερειακή πολιτική, την πολιτική της συνοχής. Εκεί είμαστε βέβαιοι ότι εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας. Στην δική μου την περιοχή, την Ακουιτανία, ε, χίλια προγράμματα ετησίως, την χάνουν χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο. Είναι αυτό επικουρικότητα. Ταυτόχρονα και εφόσον οι εθνικοί προπολογισμοί υπόκεινται σε πιέσει άνευ προηγουμένου, δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή για να εξέλθουμε από ένα σύστημα που ο κοινοτικό προπολογισμό χρηματοδοτείται από τους εθνικούς, αλλά βαρύνει τους προπολογισμού αυτού που δεν αντέχουν άλλων. Δεν αντέχουν. Θέλουμε μήπως, να, μήπως είναι μάλλον η στιγμή να επιστρέψουμε στην πρώτη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρχή που παραμένει καθαγιασμένη στις συνθήκες αρχή βάσει της οποίας οι ευρωπαϊκές δαπάνες πρέπει να χρηματοδοτούνται από τους ίδιους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ αρκετοί από εσά ανέφεραν το ζήτημα αυτό στην πρωινή συζήτηση. Το σημερινό σύστημα όπου τα κράτη-μέλη χρηματοδοτούν τον κοινοτικό προπολογισμό έχει γίνει πλέον ε, κάτι που δεν το αντέχουν. Είναι βαθιά αδικό γιατί υπάρχει μεταξύ ημών μισή, γύρω στις έξι χώρες, οι οποίες είναι ευνοημένες και πληρώνουν, συνεισφέρουν πολύ λιγότερα, σοβαρά λιγότερα από ό,τι επιτρέπει ο εθνικός τους πλούτος και θα έπρεπε να είναι η συνεισφορά τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια κάποιες χώρες αυτό το σύστημα δεν είναι ευνοημένε. Σημειώνω ότι ουδέποτε δεν βλέπουμε τα πράγματα από αυτή την πρόπτικη, ιδίω από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή στι συναντήσει των Υπουργών Οικονομικών συμβαίνει αυτό, αλλά ελπίζω οι βουλευτέ των Εθνικών Κοινοβουλίων, ιδίω των χωρών που αφορούν τα προβλήματα αυτά, θα συζητήσουν δημοσίω όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτή η διάσκεψη είναι μια ευκαιρία για να θέσουμε στου εαυτού μα αυτά τα ερωτήματα μαζί με πολλά άλλα. Επίσης, σημείωσα από την πρωινή συζήτηση, μετά από παρέμβαση του εκπροσώπου της Γαλλικής Γερουσίας, του κυρίου Μαρινή, ότι υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα. Μήπως πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ των προβλημάτων που είναι ιδιάζοντα της Ευρωζώνης και των χωρών δηλαδή των χωρών που έχουν αυτή τη στιγμή ένα κοινό νόμισμα και των υπολείπων. Θα μπορούσαμε και αυτό να το δούμε στην απογευματινή συζήτηση, αλλά μπορούμε ήδη να το έχουμε κατά νου. Εν είδη λοιπόν εισαγωγή, αυτά ήθελα να αναφέρω. Και θα ήθελα τώρα, κύριε Επίτροπε, να μας παρουσιάσετε τις αδρές γραμμές του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ερχόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Ε, ε, είναι μια βροχερή ημέρα. Ε, είναι συνηθισμένο αυτό στις Βρυξέλλες, όπως οι απεργίες. Σήμερα απεργούν οι ταξιτζίδες στις Βρυξέλλες. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρη η σημερινή συνεδρίαση μία εβδομάδα πριν την αποφασιστική ε, συνάντηση ε, των Ευρωπαίων ηγετών για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Να δούμε λοιπόν ε, ποιο είναι το όραμα για την Ευρώπη μέχρι το 2020, ποια η περικοδότηση και καλό είναι που έχουμε εκπροσώπους εκλεγμένους ο λαών από 27 χώρες. Δεν ξέρω αν πάρει βρίσκονται και Κροάτες, αλλά τα 27 κράτη-μέλη εκπροσωπούνται. Το είπε προηγουμένως και ο Λιρέν και τώρα ο Αλέν Λαμασούρ. Είναι διαφορετικό το κλίμα πλέον στην Ευρώπη και μεγάλες οι προκλήσεις. Η εξηγίαση των δημοσίων οικονομικών είναι η μητέρα όλων των πολιτικών. Όλες οι πολιτικές μας δηλαδή από το 2009 2011 δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτή τη διάσταση. Ψάχνουμε ένα μείγμα πιο ισόρροπο ε, στην οικονομία και έχει ε, λοιπόν ε, τώρα αλλάξει και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και ο Ευρωπαϊκός Υπολογισμός. Χαίρομαι λοιπόν τώρα είναι η ώρα και ο τόπος η Ευρώπη να αποδείξει τη χρησιμότητά της. Όχι στο μέλλον. Αλλαγέ θα γίνουν, ε, βέβαια, αλλά τώρα θα πρέπει να αποδείξουμε τη χρησιμότητά χρησιμότητά Και από εκεί θα κρυθούμε από το αποτέλεσμα, από τη δυνατότητα που θα έχουμε να λύσουμε την οικονομική κρίση. Και αυτό έχει σχέση και με τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, γιατί είναι διαφορετικός στη δομή του από τους ε, εθνικούς προϋπολογισμούς. Ε, ε, δεν είναι πανάκια. Έχει όμως τη δυνατότητα ως επενδυτικός προϋπολογισμός να είναι απάντηση για το πώς συνδυάζεται η εξυγίαση με την ανάγκη να βρούμε μακροπρόθεσμα χρηματοδότηση των επενδύσεων, δηλαδή για την ανταγωνιστικότητα και τις θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η προστιθέμενη αξία και εδώ έρχεται η διαφορά με τους άλλους προϋπολογισμούς. Θα το γνωρίζετε ε, ότι είναι ο μόνος πάντα ισοσκελισμένος προϋπολογισμός στον κόσμο. Δεν μπορούμε εμείς να βγούμε στις αγορές. σε αντίθεση με τους υπουργού οικονομικών των κρατών μελών ή τις τράπεζες Το μόνο που μπορούμε να δαπανίσουμε είναι αυτό που ε, εισπράττουμε ως τι εθνικέ συνεισφορές, τους δασμούς ε, και άλλες εισφορές των κρατών μελών. Για το μέλλον λοιπόν τώρα. Έχουμε κάποιες σαφείς προτάσεις που ευθυγραμμίζονται με την ανάπτυξη, με την ανταγωνιστικότητα, με τις θέσεις εργασίας. Γνωρίζουμε ότι είναι πολύ δύσκολο ε, να βρεθούν ε, εθνικοί πόροι για χρηματοδότηση, με εξαίρεση τη Σουηδία που έχει και ενσιανού τύπου ε, οικονομία και φορολογικά κίνητρα, αλλά στις υπόλοιπε χώρε, το πρώτο θύμα της λιτότητα και των οικονομιών είναι ε, τα χρήματα για τις επενδύσεις. Και επειδή δεν είναι ε, πολύ κοινωτικοποιημένα όπως άλλες μορφές δαπανών, ε, πέφτουν θύματα λοιπόν οι επενδύσεις σε αυτό το βωμό. Τι προτείνουμε λοιπόν με αυξανόμενη τα είναι λεγόμενος Horizon 2020. Είναι ε, μια νέα γενιά ερευνητικών προγραμμάτων. Για πρώτη φορά όμως στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει ε, σαφής ε, ένωση της έρευνας με την καινοτομία. Γιατί εδώ πραγματικά χωλαίνει η Ευρώπη. Έχουμε δημόσιες επενδύσεις για την έρευνα, αλλά δεν έχουμε απαραίτητο εμπορική καινοτομία, μεταφορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων, ε, όπως σημαίνει αντίστοιχα στις Ηνωμένε Πολιτείε. Από 55 δισεκατομμύρια για την έρευνα η αρχική μας πρόταση πειράσει στα 80 δις δεν ξέρω ποια θα είναι τα τελικά ποσά, αλλά αυτή ήταν η αρχική πρόταση του 2011. είναι η νέα γενιά προγραμμάτων των ερευνητικών, το λεγόμενο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και μέχρι τώρα έχουμε λάβει 95 αιτήσει για χρηματοδότηση έρευνα στο πρόγραμμα αυτό από 400 περίπου ερευνητέ είτε πρόσωπα είτε ερευνητικά ιδρύματα. 16.000 υποτροφίες έχουν δοθεί ή χρηματοδότηση σε 100.000 περίπου πρόσωπα και ερευνητικά κέντρα σε όλη την Ευρώπη και πιθανότατα, όχι πιθανότητα, είναι βέβαιο ότι είναι η πιο σημαντική πηγή χρηματοδότησης της έρευνας στην Ευρώπη. Δεν συμβαίνει αυτό σε πολλές χώρες από τον εθνικό του προπολογισμό. Έχουμε λοιπόν αυτή τη νέα γενιά προγραμμάτων, των ερευνητικών προγραμμάτων που εφαρμόζονται αυτόν τον καιρό και προτείνουμε ένα νέο είδος ε, στενότερης σχέσης στον ορίζοντα 2020, ε, είπαμε, της έρευνας με την καινοτομία. Έχουμε ένα ειδικό πρόγραμμα κόσμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αρχική πρόταση, χρηματοδότηση, αλλά νομίζω θα διατηρηθεί αυτό ε, το κονδύλι και 1,4 δις στα λεγόμενα χρηματοδοτικά μέσα που θα αποτελέσουν μοχλό ε, και εγγυήσει δηλαδή ε, και κεφάλαιο κινδύνου ε, που λείπει για την εγγύηση των επενδύσεων από την Ευρώπη και την οικονομική δυνατότητα μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έχουμε και μια νέα γενιά προγραμμάτων για την εκπαίδευση και την κινητικότητα των νέων που έχει εντοπιστεί ως μεγάλο πρόβλημα. Φαντάζομαι ο κύριος Άντορ θα σας είπε πόσο σημαντικό είναι να δώσουμε ε, και πάλι ε, μια προοπτική για το μέλλον τους νέους στην Ευρώπη. Πέρα από τα πρωτοσέλιδα που είδαμε για τον αέρασμο και το πρόβλημα χρηματοδότησης που είχε στο τέλος του 2012, έχουμε και άλλα στοιχεία και προγράμματα για τη διαβίου μάθηση και αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι η κινητικότητα των νέων στην Ευρώπη γιατί έχουμε διαφορά στην ανεργία των νέων. Ας πούμε στην Αυστρία είναι κάτω του 5% ενώ στην Ισπανία και αλλού είναι υψηλή ανεργία. Λοιπόν, η κινητικότητα είναι μια μερική απάντηση που θα μπορούσε να ενισχυθεί περισσότερο και ε, με ένα είδος ε, μαθητείας και υποτροφιών στην Ευρώπη. Πώς λοιπόν μπορούμε να κινητοποιήσουμε τα λίγα χρήματα που υπάρχουν στον κοινοτικό προπολογισμό. Αναζητούμε και πάλι μόχλευση από ένα μέσο που ονομάζεται διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη, Connecting Europe. Ε, αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα ε, διεθνή και για την πραγματική ασφάλεια, έτσι, ουσιαστική ασφάλεια. Ε, δεν είναι απλές διακηρύξεις. Χρειαζόμαστε διασύνδεση των κρατών μελών μεταξύ τους ε, σε δίκτυα. Και επίσης η ψηφιακή οικονομία είναι κάτι που δεν... Ε, υπάρχει. Έχουμε πρόβλημα στη μακροπρόθεσμη επένδυση, ιδιαίτερα στις μεταφορές, γιατί είναι μεγάλος ο κίνδυνος ο μακροπρόθεσμος. Και θα πρέπει επίσης να αναβαθμίσουμε και την αξία και την τη βαθμολογία θέλετε αυτών των προγραμμάτων με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και είναι ε, μεγάλη η μόχλευση που μπορεί να προκύψει. Τώρα έχουμε πιλωτικά λεγόμενα προγράμματα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις υποδομές μεταφορών. Αυτές είναι οι συγκεκριμένες θέσεις του προεπολογισμού ε, ε, που αφιερώνονται σε ένα κλάδο ή αποτελούν μοχλό. Ε, οι μεγαλύτερες δαπάνες ε, ε, αφιερώνονται στη συνοχή και στην ανάπτυξη της υπαίθρου και αυτό είναι και μια ευκαιρία επαναπροσανατολισμού των δαπανών προς τις θέσεις εργασίας, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Πώς γίνεται αυτό? Με λεγόμενες συμβάσεις εταιρικής σχέσης Υπάρχει η μακροοικονομική αιρεσιμότητα εκ των προτέρων για τις δαπάνες, συνδέονται με κάποιες προποθέσεις. Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλές σήμερα στην Ευρώπη και στις χώρες μας. Αν δείτε όμως ποιοι είναι οι στόχοι και πόσο στενή είναι η στόχη για τις πιο πλούσιες περιοχές στην Ευρώπη, ε, καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να δαπανούμε περισσότερα για την ανταγωνιστικότητα, για την καινοτομία. Ε, το θέμα είναι αυτό λοιπόν, πώς η ε, ανάπτυξη πέθρου ή η ε, συνοχή ε, και οι άμεσες πληρωμές προς τους αγρότες, πώς θα επαναπροσανατολιστούν και θα διοχετευθούν προς τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Είμαστε λοιπόν μια εβδομάδα πριν τη Σύνοδο. Η πρώτη του Νοεμβρίου δεν επέτυχε, αλλά δεν ήταν μια χαμένη ευκαιρία. Προχωρήσαμε, γνωρίζουμε περισσότερο τώρα για το ποιες είναι οι αδιαπραγμάτευτες θέσεις των κρατών, ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές όπως λέμε ε, και αυτό ε, βοήθησε σε προετοιμασία ε, για να μην αβαγήσει και η δεύτερη προσπάθεια, η δεύτερη σύνοδος της 7ης και 8ης Φεβρουαρίου Για πρώτη φορά στην ιστορία της ευρωπαϊκής οικοδόμησης θα μπορούσε ε, ε, ο δανεισμός να είναι μικρότερος. Ο κύριος Φαν ε, Ρομπέι έκανε μια πρόταση για λιγότερα, 20 ε, δισεκατομμύρια λιγότερα ε, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Χρειάζεται βέβαια και ειδική πλειοψηφία. Βλέπω σήμερα στην εφημερίδα Frankfurter Allgemeine μια ωραία συμμαχία εδώ ε, Γερμανούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Άλβαρο πρώτος, ε, είναι ευρεία η συμμετοχή, λέει η κυρία Χάουκ, ε, Τσέντεου, Γιούτα Χάουκ από τους σοσιαλιστές, ο κύριος Άλβαρο, η κυρία Τρίπελ από τους Πρασίνους. Είναι μια ευρεία ε, συμμαχία, ευρύ το φάσμα των Γερμανών βουλευτών που είναι ενωμένοι εδώ για να αντιπροσωπεύσουν, για, να υπερασπιστούν τον κοινοτικό προϋπολογισμό και η αξία του ποια είναι, οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις και επίσης η προβλεψιμότητα των επενδύσεων. Έτσι είναι η φύση της χρηματοδότησης από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Είναι πολυετή τα προγράμματα και ε, η βάση είναι πάντα η σταθερότητα. Δυστυχώς τη λογική των διαπραγματεύσεων πριτανεύει η ε, εθνική θεώρηση κάθε φορά και ο καθένας θέλει να εξασφαλίσει τα κεκτημένα του. Αντί να ε, κοιτάμε προς το μέλλον. Η γενική συντηρητική θέση των κρατών μελών είναι να υπερασπίζονται την ε, γεωργία και τις άμεσες ενισχύσεις στη γεωργία. Θα πρέπει όμως να εξυγχρονιστεί ο προϋπολογισμός και επίσης πολύ... Ε, καλά γνωρίζω ότι ο παρακαθήμενος, ο πρόεδρος, θα μιλήσει για τη γεωργία και πόσο σημαντική είναι αυτή και για την Ιρλανδία. Ναι, και για το κοινοβούλιο αυτό που έχει σημασία είναι η απλούστευση, αλλά αυτό είναι και οι κανόνε του παιχνιδιού για το πώ θα δαπανώνται τα κονδύλια. Ο λεγόμενος νέος δημοσιονομικός κανονισμός ζητούν δραματικά απλούστευση, μείωση τη γραφειοκρατίας οι ενδιαφερόμενοι και θα πρέπει να είναι από τους στόχους μας, οπωσδήποτε και υψηλή προτεραιότητα ε, την ερχόμενη περίοδο. Και επίσης θα πρέπει να εντοπίσουμε ε, λεγόμενα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα, γιατί ό,τι προσπάθεια και να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα χρειαστεί στο μέλλον να χρηματοδοτηθεί περισσότερη Ευρώπη, συν την Κροατία που θα έρθει να προσθεθεί ως 28 ε, κράτος και περισσότερες εξουσίες. Περισσότερη Ευρώπη για πρώτη φορά με ίσως λιγότερα χρήματα από ό,τι είχαμε τώρα. Γι' αυτό θα χρειαστεί η μόχλευση και άλλα χρηματοδοτικά μέσα. Ε, με χαρά λοιπόν περιμένω τη συζήτηση. Δεν ξέρω αν σας έπεισα. Σας ευχαριστώ και πάλι για την ευκαιρία που μου δώσατε να ε, απευθυνθώ σε εκλεγμένους ρετούς εκπροσώπους λαών. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πίτροπε, κύριε Πρόεδρε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σε απευθύνω τον λόγο σήμερα και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Επίτροπο για την αρχή του ομιλία, στην οποία προσίασε κάποια ζητήματα τα οποία θα αναφέρω και εγώ στη δική μου ομιλία σήμερα. Αγαπητοί συνάδελφοι, το κυριότερο θέμα τη Ιρλανδική Προεδρίας είναι η ανάπτυξη και η σταθερότητα. Η διασφάλιση τη σταθερότητα, η οποία θα διασφαλίσει τις θέσει εργασία και την ανάπτυξη. Για αυτό το σκοπό χρειάζεται να οικοδομήσουμε μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία ευέλικτη στι καλέ εποχέ και βιώσιμη στις κακέ. Χρειαζόμαστε σταθερό ευρωπαϊκό κλίμα όπου τα κράτη-μέλη θα αλληλοϊποστηρίζονται κατά των αρνητικών οικονομικών δυνάμεων και όχι βάσει ανταγωνισμού μεταξύ του και συμφέροντος μόνο μιας χώρας. Η Ευρώπη είναι ισχυρότερη, ενωμένη και σε αυτό το δύσκολο οικονομικό κλίμα αυτή η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαίων είναι σημαντικότερη από ποτέ. Το λογότυπο της Ευρώπης είναι ενωμένη στη διαφορετικότητα και πρέπει να αντικατοπτρίζουμε αυτή την αρχή για να συνεχίσουμε ως ανταγωνιστές σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο υπήρξε μια σημαντική εξέλιξη για τη διασφάλιση της καθοδήγησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τα κράτη-μέλη για το σχηματισμό δημοσιονομικής πολιτικής πριν ξεκινήσει η διαδικασία διαρθρωτικού προϋπολογισμού και για την ενίσχυση της επιτήρησης και της ολοκλήρωσης χρειάζεται επαγρύπνηση σε εθνικό επίπεδο και χρειάζεται τα Εθνικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχουν δημοκρατική λογοδοσία και υπευθυνότητα η Ιρλανδική Προεδρία έχει αναλάβει τη δέσμευση και έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της. Είναι σημαντική, είναι ζωτική σημασία σε αυτή η διαδικασία, διότι θέτει υπό εξέταση τι πολιτικέ των κρατών μελών. Παρακολουθεί και ελέγχει τις προτεραιότητε δαπανών, ώστε να είναι βέβαιοι ότι κάνουν σωστέ επιλογέ στα κράτη-μέλη. Ωστόσο, αποτελεί μια ευκαιρία μια ευκαιρία να διασφαλιστεί ότι η έρευνα, η καινοτομία και η ανάπτυξη έχουν ενσωματωθεί στις εθνικές πολιτικές. Σε όλη την ιστορία οι κοινωνίες ε, έδιναν μεγαλύτερη σημασία στις προτεραιότητες που άρμοζαν στη συγκεκριμένη εποχή. Σήμερα αυτή η προτεραιότητα είναι η καινοτομία. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη της πρόκληση και ε, ως το 2050 θα έχει μόλις 6% του παγκόσμιου πληθυσμού οι σημαντικοί παίκτες παγκοσμίω ε, ε, έχουν να αντιμετωπίσουν τις αναδυόμενες δυνάμεις, την Κίνα, την Ινδία, τη Βραζιλία. Σε αυτό το οικονομικό κλίμα πρέπει οπωσδήποτε να αδράξουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε ώστε να επιτύχουμε την καινοτομία μέσω όλων των εθνικών προπολογισμών. το, η αρχική πρόταση πολιετού δημοσιονομικού σχεδίου ε, της Ευρώπης κατά την ελλανδική άψη έχει επιτύχει τη σωστή ισορροπία. Επικυρώνουμε ε, και τις μειώσεις και ε, την, τον έλεγχο των δαπανών. Θεωρούμε ότι το κλίμα, το οικονομικό κλίμα είναι δύσκολο και πολλά κράτη-μέλη μεταξύ των οποίων και η Ιρλανδία υποφέρουν από τις επιπτώσεις της παγκόσμια κρίσης. Αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να κάνουμε σπασμωδικές αντιδράσεις που θα θέσουν σε κίνδυνο τη δουλειά των προηγούμενων δεκαετιών. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε το μέλλον της Ευρώπης και των πολιτών της. Η Ιρλανδία αποτελεί το παράδειγμα χώρας που επιτυχώς αξιοποίησε τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ενισχύσει τις δυνατότητες της επενδύοντας σε υποδομές και σε ανθρώπινο δυναμικό. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες επαναδιοργανώσαμε την οικονομία μας ώστε να μπορούμε να επενδύουμε περισσότερο σε τομείς γνώσης της οικονομίας μας. Αυτό θα αντικατοπτρίζεται ως στοιχείο κλειδί της Ελληνικής Προεδρίας. Εμείς θα διασφαλίσουμε ότι τα ε, χρηματοοικονομικά προγράμματα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υποστηρίξουν την καινοτομία και την ανάπτυξη βασικών υποδομών για την ανάπτυξη η Ιρλανδική θέση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο έχει δύο πτυχές. Πρέπει να διασφαλίσουμε τον προπολογισμό μέσω ίδιων πόρων και δεύτερον θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τις δαπάνες στην αγροτική πολιτική. Τα διαρθρωτικά ταμεία μόνο 6% αντιπροσωπεύουν η Ιρλανδία θα χρειαστεί να διατηρήσει ουδέτερη θέση κατά την ε, διαπραγματεύσεις στη διάρκεια της Προεδρίας ως ε, υπεύθυνη πολιτικής έχουμε την ευθύνη να ζητήσουμε βοήθεια για να μπορέσουμε να χαράξουμε τις πολιτικές. Εγώ θεωρώ ότι ένα από τα στοιχεία κλειδιά θα είναι να δώσουμε περισσότερη σημασία στην έρευνα και στην καινοτομία. Ο πίνακα αποτελεσμάτων τη Ευρωπαϊκή Καινοτομία, το EIS, είναι μια συγκριτική ε, αξιολόγηση της καινοτομία στα διάφορα κράτη-μέλη. Το EIS 2007 περιλαμβάνει δείκτες καινοτομία και αναλύσεις τάσεων για τα 27 κράτη-μέλη και άλλα. Οι κύριοι ανταγωνιστές της Ευρώπης, όπως Αυστραλία, Βραζιλία, Κίνα, Ινδία, Νότια Αφρική, Καναδά, Αφρική και Ηνωμένε Πολιτείε. Οι επιδόσεις καινοτομία στις ΗΠΑ Πολιτείες, ε, στην Νότια Κορέα και στην Ιαπωνία είναι πάνω του συνόλου των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε πίσω. Είμαστε πίσω σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην παγκόσμια σκηνή πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα και να δώσουμε, να θέσουμε την καινοτομία στο επίκεντρο. Το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη θα αποτελέσουν τα κύρια εργαλεία για την υποστήριξη της έρευνας, της ανάπτυξης για τις επιστήμες, την τεχνολογία, όπως ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Επίτροπος. Ωστόσο, δεν υπάρχουν εθνικά προγράμματα, ακόμη τα προγράμματα αξιολογούνται από πάνελ ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων. Δεν υπάρχει λοιπόν δημοσιονομικός στόχος. Έχουμε έναν εσωτερικό ανταγωνισμό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ιρλανδία συμμετείχε ιδιαίτερα στις αιτήσει ε, χωρίσεις ε, κονδυλίων για το πρόγραμμα πλαίσιο μέχρι το έχουμε υποβάλει πάνω από 6.000 αιτήσει για τη συμμετοχή στο FP7. Ω αποτέλεσμα, ένας μεγάλος αριθμός ετούντων ε, πέτυχαν τις προτάσεις με ποσοστό επιτυχίας άνω του 23% με ε, ε, χρηματοδότηση άνω των 438 εκατομμύριων ευρώ. Η Ιρλανδία έχει εξαιρετικέ επιδόσει στα μικρή και μεσαίας κλίμακας έργα και η τάση συνεχίζεται με διασφάλιση 40% τη χρηματοδότηση αυτή σε μικρή και μεσαίας κλίμακας έργα. Το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την κοινοτομία βοηθά στη συμμετοχή μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που βρίσκονται στη καρδιά του 98% της επιχειρησιακής δραστηριότητας στην Ευρώπη αποτελούν παράγοντα κλειδί για την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας στο Horizon 2020 θα αυξήσει τη συμμετοχή των ΜΜΕ από 15% σε 20%. Το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο χρηματοδότησε για παράδειγμα στην Ιρλανδία 3.000 θέσεις εργασίας από το 2007 και όπως είπα το 23% της Ιρλανδίας είναι άνω του μεσόρου της ε, Ευρώπης. Για να συνεχίσουμε να δημιουργούμε θέσεις εργασίας και να τονώνουμε την οικονομία πρέπει να προωθούμε τη συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα. Το προτινόμενο ορίζοντα 2020 πρέπει να επιτύχει αυτό το στόχο. Θα πρέπει να δημιουργήσει ένα σύστημα που θα υποστηρίζει την ευρωπαϊκή ηγεσία, τη βιομηχανική ανάπτυξη και θα αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Το Horizon 2020 είναι οικοδομένο σε τρεις ε, πυλώνες επιστήμη, βιομηχανία και κοινωνικές προκλήσεις. Προτεραιότητα κατά τη δική μας προεδρία, προεδρία είναι η πρόθεση των πρωτοβουλειών κατά πολέμησης της ανεργίας και ειδικότερα της απασχόλησης των νέων. Τα προγράμματα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αποδείξει ότι δημιουργούν θέσεις εργασίας και πρέπει να συνεχίσουμε την υποστήριξη προς αυτά τα προγράμματα. Η Ιρλανδική Προεδρία αναγνωρίζει τη σημασία της έρευνας ως εργαλείο όπου ερευνητές, η τεχνολογία και η καινοτομία μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Εφόσον υλοποιηθεί, θα βελτιώσει τις επιδόσεις της Ευρώπης στην έρευνα. Θα ήθελα να εστιάσουμε την προσοχή μας σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα που αφορά την Ιρλανδική Προεδρία όσον αφορά την καινοτομία, δηλαδή της άδειας ευρεσιτεχνίας. Η επίσημη υιοθέτηση του σχετικού κανονισμού από το Συμβούλιο έλαβε χώρα υπό την Κυπριακή Προεδρία και η Ιρλανδική Προεδρία θα, προετοιμαστεί, θα προετοιμάσει τα κράτη-μέλη για την επίσημη υπογραφή στο πρώτο μισό του 2013. Αυτή η πρωτοβουλία θα βοηθήσει όσους καινοτομούν να προστατεύουν τις ε, επινοήσεις τους, τα επινοήματά τους. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα υποφεληθούν από το μειωμένο κόστος και η προστασία που απορρέει από αυτόν τον κανονισμό θα βοηθήσει όσους καινοτομούν. Αυτό αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Για να επανέλθουμε στο ζήτημα της απασχόλησης των νέων, η επίλυση αυτού του ζητήματος που έχει φτάσει η ενεργεία στο 40% σε ορισμένα κράτη-μέλη θα αποτελέσει θεμέλιο λίθο της Ιρλανδικής Προεδρίας Πιστεύω ότι οι νέοι είναι στην καρδιά τη ε, μεταμόρφωση τη Ευρώπη προ τι νέε τεχνολογίε. Πρέπει να ενθαρρύνουμε του νέου ανθρώπου στην αγορά εργασία να χρησιμοποιούν τι δεξιότητέ του. Πρέπει να του προσφέρουμε ένα καλύτερο μέλλον. Σε αυτέ τι δύσκολε εποχέ υπάρχουν ευκαιρίε καινοτομία και αλλαγή. Πρέπει να εμπιστευτούμε του νέου, να του παρέχουμε τα εργαλεία να τους ενθαρρύνουμε να καινοτομούν και να φέρουν την Ευρώπη μπροστά οι χώρες με ισχυρά ρυθμιστικά περιβάλλοντα, με ανεπτυγμένες υποδομές, χώρες όπου γίνονται σημαντικές επενδύσεις και έρευνα και με πολλά ταλέντα θα αποτελέσουν πυρήνες ανάπτυξης. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνεργαστούν ώστε να θέσουν την καινοτομία στο επίκεντρο των δημοσιονομικών τους πολιτικών. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου έτσι θα βγούμε από την καταιγίδα και θα καταλήξουμε σε μια πιο ισχυρή ένωση, καινοτόμο ένωση γεμάτη γνώση. Για να ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρο, 28 και 29 Απριλίου φέτος η σχετική επιτροπή της Ελλανδικής Προεδρίας θα συναντηθεί με εκπροσώπους των Επιτροπών Απασχόλησης και Νέων των 27 χρόνων μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κυρία θέματα ζήτηση αυτής της συνεδρίας θα είναι στρατηγικές καταπολέμησης της ανεργίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα θέματα του Horizon 2020. Βάσει αυτού του προγράμματο, το Ελλανδικό Κοινοβούλιο θέτει στο επίκεντρο την έρευνα και την καινοτομία για τη δημιουργία θέσεων εργασία και ανάπτυξη. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με του ομολόγου μα από όλη την Ευρώπη. Η κρίση αποτελεί κίνητρο. Όχι απλό, αλλά είναι πιστευτό. Η εμπειρία μας λέει ότι η ανάκαμψη θα εξαρτηθεί από τις δράσεις σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, από την υλοποίηση. Εμείς είμαστε περήφανα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και 40 χρόνια. υπομονούμε να συνεχίσουμε τα επόμενα 40 χρόνια συνεργαζόμενοι για την ειρήνη, τη σταθερότητα, την ευμερία στο μέλλον της Ευρώπης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ε, για το μήνυμα αυτό ε, για τη μεγάλη εμβέλεια της Ιρλανδικής Προεδρίας. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον η εισηγήτριά μας, την Άνια Ενσεν, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι από τη Δανία φιλελεύθερη ε, και παρακαλώ τους υπολείπους ομιλητές να περιοριστούν όσο γίνεται χρονικά γιατί έχουμε καθυστερήσει για να γίνει μια ουσιαστική ανταλλαγή. Παρακαλώ, Αν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να εξηγήσω την κατάσταση σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2014 και πώς το βλέπουμε αυτό στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Το πρώτο πρόβλημα φυσικά είναι ότι δεν έχουμε ακόμα πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δεν ξέρουμε πώς θα χειριστούμε τη νομική βάση και το αν ε, θα κολλήσουμε σε μια κατάσταση χωρίς ε, λύση, αλλά θα δούμε τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Αλλά, όπως ανέφερε ο κύριος Λεβαντόσκι, επιτάπητος ε, Υπάρχει μια πρόταση που θα αγώσει τον προϋπολογισμό στα επίπεδα του 2008 μέχρι το 2020. Για τα επόμενα 7 χρόνια δηλαδή θα έχουμε προϋπολογισμό στο επίπεδα, στα επίπεδα του 2008, δηλαδή 5% λιγότερο από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα. Οι περικοπές θα αφορούν και τον γεωργικό τομέα, ε, λέω εγώ προσωπικά, μπορεί άλλοι να έχουν άλλη άποψη. Ε, θα έχουμε περικοπές όσον αφορά την συνοχή και θα υπάρχει από ό,τι φαίνεται αύξηση των δαπανών για την έρευνα, την υποδομή των μεταφορών. Μάλλον όχι όμως στο βαθμό που είδαμε στην πρόταση της Επιτροπής που ήταν πρόταση που βρίσκει ισχυρή υποστήριξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα δούμε πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα, αλλά ο φόβος του Κοινοβούλιο είναι ότι όχι μόνο θα έχουμε έναν ε, πολύ λίγο φιλόδοξο προϋπολογισμό ως προς τα ποσά, αλλά και με πολύ λίγη ευελιξία, ώστε να μην μπορούν να αλλάξουν οι προτεραιότητες από τώρα μέχρι το 2020. Και θα ήθελα να σας θυμίσω ότι την τελευταία φορά θέσαμε πολιετές πλαίσιο υπό την προεδρία του ε, Τόνι Πλέρ, ε, το οποίο αποτέλεσε αργότερα από κείμενο διαπραγμάτευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, αλλά μισό χρόνο μετά έκλεισαν οι Ρώσοι την παροχή του αερίου προς τη Βουλγαρία και σκεφτήκαμε ότι ούψ, χρειαζόμαστε μια ενεργειακή πολιτική, δεν έχουμε όμως τα λεφτά για αυτήν. Ευτυχώς υπάρχει περιθώριο στην είχαμε κάποιο περιθώριο στον προπολογισμό τη Γεωργία, οπότε μπορέσαμε να βρούμε τα χρήματα, αλλά είμαι αρκετά σίγουρη ότι δεν θα έχουμε τόση ευελιξία την επόμενη φορά. Χρειαζόμαστε λοιπόν την, την ευελιξία λόγω των αλλαγών που μπορεί να υπάρξουν στον κόσμο από τώρα μέχρι το 2020. Νομίζω ότι θα μπορούμε να είμαστε αρκετά βέβαιοι ότι θα προκύψουν νέε καταστάσει. Σημαντικό είναι ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συζητήσει τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό με, τα Εθνικά Κοινοβούλια για διάφορου λόγου, μερικοί από του οποίου ήδη αναφέρθηκαν. Ο προπολογισμό Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μικρό, είναι όμω προπολογισμό επενδύσεων και για πολλά κράτη-μέλη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλά κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται στην κατάσταση όπου ο ευρωπαϊκό προπολογισμό στηρίζει το 70% των δημοσίων επενδύσεων του. Για κάποια κράτη-μέλη λοιπόν είναι ζωτική σημασία. Επίση έχουμε την έρευνα και άλλα πράγματα, άλλου τομεί τομείς στους οποίους συνεργαζόμαστε και δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε το επίπεδο που φτάνουμε εάν δεν συνεργαζόμασταν. Και σημειώνω ιδιαίτερα την ομιλία της Ιρλανδικής Προεδρίας που τονίζει ότι για μια μικρή χώρα ε, είναι πολύ ζωτικό το θέμα αυτό. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συχνά μιλάμε για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και σίγουρα μπορούμε να κάνουμε μαζί πράγματα που δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε μόνοι μας. Θα πρέπει να το συνειδητοποιούμε αυτό και γι' αυτό θα πρέπει ε, εκεί να καταβάλουμε σημαντικές προσπάθειες. Και να συνδυάσουμε τις προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης μπορεί να βρούμε τομείς όπου, όπου ο προπολογισμό Ευρωπαϊκής Ένωση μπορεί να βοηθήσει στην ε, δημοσιονομική εξυγίανση στα κράτη-μέλη. Στη δική μου χώρα, τη Δανία, ε, έχουμε περικόψει τις δαπάνες για την εξωτερική πολιτική, διότι έχουμε τώρα την κοινή εξωτερική πολιτική. Μπορούμε λοιπόν με τη συνεργασία να εξοικονομήσουμε χρήματα στις πατρίδες μας. Και υπάρχουν τομείς που σχετίζονται με τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, όπου μπορούμε να μειώσουμε το εθνικό κόστος, να κάνουμε τα πράγματα με πιο φθηνό τρόπο, εφόσον τα κάνουμε μαζί. Και αυτά θα πρέπει να συζητήσουμε εδώ. Ποιοι είναι οι τομείς όπου τα... μπορεί να υπάρξουν περικοπές στους εθνικούς προϋπολογισμούς ε, λόγω της συνεργασίας μας γενικά. θα πρέπει να πούμε ότι δεν θα πρέπει να θεωρούμε τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό μόνο προϋπολογισμό δαπανών. Είναι προϋπολογισμός, ε, είναι και προϋπολογισμός εξοικονόμησης και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η επικεφαλίδα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον προπολογισμό τη επόμενη χρονιά είναι η ανάπτυξη. Θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε αρκετά ε, ε, χρήματα ε, για να επενδύσουμε, διότι ιδιαίτερα το θέμα τη ενεργεία των νέων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει λοιπόν να βάλουμε στην άκρη κάποια χρήματα και να βρούμε και σε εθνικό επίπεδο χρήματα για τα νέα αυτά προγράμματα που επιτρέπουν στου νέου ανθρώπου να μπουν στην αγορά εργασία. Υπάρχουν κράτη-μέλη όπου οι δημογραφικέ εξελίξει σημαίνουν ότι σε λίγα χρόνια ε, δεν θα υπάρχει επαρκές ε, εργατικό δυναμικό. Και θα έχουμε μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων ε, που δεν κατάφεραν να μπουν στην αγορά εργασίας. Αυτά λοιπόν θα είναι πολύ σημαντικά για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και μια τελευταία παρατήρηση, αλλά πρέπει να την πω τώρα που έχουμε εδώ τους εθνικούς βουλευτές. Έχουμε ένα πρόβλημα με τους οικονομικών σα επειδή ε, δεν θέλουν να υπογράψουν ε, την επιταγή που υποσχέθηκαν. Αυτό είναι αυξανόμενο πρόβλημα και θα είναι πρόβλημα μεταξύ των κρατών μελών, διότι τα κράτη-μέλη που έχουν να πληρώσουν λογαριασμούς από τα διαστατικά ταμεία δεν θα λάβουν εγκαίρως τα χρήματά τους. Από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα υπερασπιστούμε ε, στεναρά τα κοινά σημεία του προϋπολογισμού. Αλλά υπάρχουν κράτη που πρέπει να λάβουν χρήματα από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ε, διότι τα χρωστάνε αλλού. Ε, εάν λοιπόν η Ισπανία, η Ιταλία, η Ιρλανδία δεν λάβουν τα χρήματα τους εγκαίρως, θα πρέπει εσείς να αντιδράσετε αντί να κρύβεστε πίσω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είναι λοιπόν μόνο θέμα χρημάτων, είναι και θέμα Ευρωπαϊκής Επιτροπής που να μπορεί να πληρεί τα καθήκοντά της ε, σύμφωνα με τους νόμους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Αν. Το λόγο τώρα έχει ο Πρόεδρος Καμπίτα από την Πορτογαλική Βουλή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή η διακοινοβουλευτική διάσκεψη συμβάλλει στο να μειώσουμε δύο σημαντικά ελλείμματα της τελευταίας διετίας στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της κρίσης. Έλλειμμα δημοκρατικής διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων και έλλειμμα συντονισμού των οικονομικών πολιτικών. Είναι άλλωστε εύγλωτο ότι το θέμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου φέτος θα είναι απασχόληση και ανάπτυξη. Αυτό αποδεικνύει ότι η αντίδραση της Ευρώπης την τελευταία διετία ήταν πάντοτε καθυστερημένη και τουλάχιστον αναγνωρίζεται στις ε, προτεραιότητες για φέτος, αλλά οι εκτιμήσεις για το 2013 δείχνουν ότι η Ευρώπη θα παραμείνει σε ύφεση. Ξεκινήσαμε από μία κρίση κρατικών χρεών. Ένα θέμα των ε, οικονομιών των περιφερειακών χωρών. Εδώ βρέθηκε μια ενιαία λύση, πολιτική λιτότητας. Όλα αυτά είχαν ως συνέπεια την συστημική διόγκωση της κρίσης, ώστε να πλήξει ολόκληρη την Ευρωζώνη και ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι αυξήθηκαν οι διαστάσεις της και η απόκριση που έδωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιτρέπει επιτέλους να αντιστραφεί αυτή η τάση. Το παράδειγμα της Πορτογαλίας είναι χαρακτηριστικό. Η Πορτογαλία συχνά αναφέρεται ως ένα παράδειγμα αποτελεσματικότητας, αποφασιστικότητας με μεγάλη εσωτερική κοινωνική συνένεση στην εφαρμογή αυστηρών πολιτικών δημοσιονομικής εξυγίανσης. Τις θεωρήσαμε απαραίτητες, όμως οι συνέπειες σε οικονομικό επίπεδο είναι καταστροφικές. Αυξημένη ανεργία, τρίτη χρονιά συνεχόμενης ύφεσης και έντονη κοινωνική κρίση. Η απάντηση πρέπει να βρεθεί και σε εθνικό επίπεδο, αλλά εδώ μας ενδιαφέρει η ευρωπαϊκή διάσταση. Γι' αυτό η στρατηγική του 2020 χαράζει έναν δρόμο, την αρχή ενός δρόμου, όπως η έμφαση στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Χρειάζονται δημόσιες επενδύσεις σε τομείς όπως εποδομές που να επιτρέψουν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την ανάπτυξη. Αυτό μας παραπέμπει σε κάτι που αναφερόταν στο προηγούμενο συζήτηση της συζήτησης, την στρατηγική για την ανάπτυξη δηλαδή, σε αυτή τη χρονική συγκυρία, αλλά στην ουσία, στο πώς θα διαρθρώσουμε την προσαρμογή των προγραμμάτων μεταρρύθμισης στην ανάγκη να αποφύγουμε δομικά διαρθρωτικά προβλήματα που να δημιουργήσουν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προβλήματα στην ε, υγιή οικονομική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Εδώ χρειάζεται μια στρατηγική όπου η υλοποίηση της προσαρμογής να συνδυάζεται με την τόνωση της ε, ανάπτυξης και της απασχόλησης, με ένα σημαντικό ρόλο των ε, κρατικών επενδύσεων δεν μπορεί να είναι η απάντηση οι περικοπές στον κοινοτικό προπολογισμό. Η απόκριση είναι περισσότερο συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών, περισσότερη δημοκρατική διαφάνεια, περισσότερη αλληλεγγύη. Δεν θα βρεθεί λύση από τη, λιγότερη, από τη μείωση και την λιγότερη Ευρώπη, αλλά από την περισσότερη Ευρώπη και την τόνωση της στρατηγικής για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Πρόεδρε. Λοιπόν, από τη Βουλή των Ελλήνων, το λόγο έχει ο κύριος Σάκη Γεροντόπουλος, παρακαλώ. Δεν επιθυμεί να μιλήσει, μάλιστα. Τότε θα δώσω το λόγο στην κυρία Χέλγα Τρίπελ. Γερμανίδα πράσινη ευρωβουλευτή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε πολύ. Τώρα εγώ θα ήθελα να μπω στο στρατηγικό ζήτημα και ερώτημα. Αφού ακούσαμε τόσο πολύ ότι χρειαζόμαστε νέα ανάπτυξη και νέες θέσει απασχόληση. Αυτό δεν το αμφισβητεί ουδής εδώ παρόν. Πότε όμως θα έρθει νέα ανάπτυξη. Κατά την άποψή μου μπορεί να έρθει μόνο αν είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε περισσότερα κατά τη ανεργία των νέων, να επενδύσουμε στην έρευνα και στην παιδεία. Αλλά εντάξει, καλή ανάπτυξη θα πρέπει να είναι όμω αηφόρο και φιλική προ το περιβάλλον για να προστατεύσουμε και το κλίμα μα. Λοιπόν, τι πιστεύω, οι επενδύσει σε παραγωγικέ γραμμέ, με οικολογική ευθύνη, με μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα ή δυνατόν και με μηδενικές εκπομπές ε, είναι οι τομείς που θα μας δώσουν ανάπτυξη. Γι' αυτό και ένας ευρωπαϊκός προϋπολογισμός που μας καθιστά σε θέση ακριβώς εκεί να επενδύουμε ε, είναι η σωστή απάντηση στην κρίση. Κατά την άποψή μου τώρα όμως η απειλή είναι να πάμε στην αντίθετη κατεύθυνση. Εάν ε, πέσει μια περικοπή 10% και ταυτόχρονα επιβληθούν και τα συμφέροντα της γεωργίας και των διαρθωτικών ταμείων, ε, και επιβληθούν και οι πλούσιες χώρες, τότε μειώνουμε την επένδυση στην έρευνα, στην ανάπτυξη και στην αηφορία που τόσο πολύ πρεσβεύουμε. Δηλαδή ε, κινδυνεύουμε ε, όλοι αυτοί οι μεγάλοι πολιτικοί λυρισμοί να πέσουν στο κενό και να ακολουθήσουμε την αντίθετη πολιτική. Θα πρέπει τώρα και με τους Ιρλανδούς στην Προεδρία να καθίσουμε και πάλι να σκεφτούμε πώς θα επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους και πώς θα τους υλοποιήσουμε. Δεύτερη παρατήρηση. στο Βερολίνο στο ΙΝΕΣ 5 ο Bill Gates και ζήτησε ένα φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ε, στη γραμμή ε, του, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στα κράτη-μέλη ακόμα διαπληκτιζόμαστε είναι σωστό ή λάθος. Ποια είναι τα κράτη-μέλη που ε, είναι τώρα πρόθυμα 11 να εισαγάγουν αυτό το φόρο. Το θεωρώ σημαντικό για τη ρύθμιση των τραπεζών και για την κατάλληλη ρύθμιση των χρηματαγορών και ταυτόχρονα θα πρέπει αυτό το κονδύλι, αυτοί οι πόροι να μπουν στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Ο κύριος Λεβαντόφσκι κατά την άποψή μου έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή πρόταση. Γιατί εάν έχουμε ίδιο πόρο αυτό το φόρο, τότε ε, οι συνεισφορές ε, του ΑΕΠ των κρατών μπορούν ε, να μειωθούν κατά το αντίστοιχο ποσοστό και έτσι κερδίζουν όλοι. Παρακαλώ το Συμβούλιο να ασχοληθεί και πάλι με το πρόβλημα αυτό και ελπίζω να μεταπιστεί κιόλας. Και μια τελευταία παρατήρηση, γιατί έχουμε τους πολλούς εθνικούς βουλευτές εδώ. Γνωρίζω τις ε, συζητήσεις σε εθνικό επίπεδο. Θέλω να τονίσω πάρα πολύ ότι αν ζητούμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηλότερο προπολογισμό, δεν το κάνουμε για λόγους μεροληπτικούς, εγωιστικού, θεσμικού συμφέροντος, αλλά γιατί θέλουμε μέχρι το 2020 να κάνουμε μια καλύτερη πολιτική για τους πολίτες της Ένωσης. Και είναι σημαντικό αυτό να το καταλάβει και το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω τώρα το λόγο για το 20 Κάμερ, το ανωσώμα του Κοινοβουλίου των Κατοχωρών στην κυρία Λόκας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στα αγγλικά. Η ε, ε, Ολλανδική Βουλή υποστηρίζει πολύ ε, ένα πιο σύγχρονο προεπολογισμό της Ένωσης, αύξηση στην έρευνα και στην ανάπτυξη και μείωση στις δαπάνες για τη γεωργία, στις επιδοτήσεις και την συνοχή. μόνο με μια ανοιχτή αγορά, με έρευνα και ανάπτυξη θα επιτρέψουμε στους ερευνητές και στις επιχειρήσεις να προοδεύσουν να βρουν νέες αγορές και νέα προϊόντα. Ε, θα πρέπει να έχουμε καινοτόμε λύσεις για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Ο εξυγχρονισμός του κοινοτικού προϋπολογισμού είναι σημαντικό βήμα προς το μέλλον. Ελπίζουμε η συζήτηση το Φεβρουάριο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να οδηγήσει ε, σε μια καμπή στον τομέα αυτό ορίζον 2020 μας βρίσκει σύμφωνος αλλά θα πρέπει να είναι ποιοτική έρευνα και ανταγωνισμός θα πρέπει να δίνουμε τα χρήματά μας στις καλύτερες ερευνητικές ε, ομάδες για να προοδεύει η έρευνα και να υποφεληθούμε όλοι τα χρήματα του ορίζοντα 2020 θα πρέπει να δοθούν σε γυναίκες ερευνήτριες ε, σε προβληματικούς τομείς στα κράτη-μέλη Ελπίζω η Ιρλανδική Προεδρία να δώσει προτεραιότητα στην ε, ενίσχυση ε, του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Τεχνίας. Ε, είναι σημαντικό για να μειωθεί η περιττή γραφειοκρατία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε λίγο βορειότερα και θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπο Μπέρναντσον από τη Σουηδική Βούλη. Καλά το είπα. Ε, Πού είστε, γιατί δεν σας βλέπω. Να, εδώ είμαι. Λοιπόν, το θέμα που ε, μας απασχολεί εδώ είναι το εξής. Πώς μπορεί ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός να βοηθήσει τα κράτη-μέλη για να βγούμε από την κρίση πώς μπορούμε να φτάσουμε στους στόχους που έχουμε θέσει. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό μπορεί να μας βοηθήσει ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός για να βγούμε από την κρίση μας. Πώς απαντούμε σε αυτό το ερώτημα. Ακούσαμε προηγουμένως. Ο κοινοτικό προϋπολογισμός θα πρέπει να εξυγχρονιστεί. Μόλις το ακούσαμε και ε, αυτή είναι η απάντηση και με τρόπο πάρα πολύ συνειδητό να επενδύουμε στα έργα που δημιουργούν εργασία, θέσεις εργασίας, δηλαδή εκπαίδευση και κατάρτιση. Είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε εκεί τη προτεραιότητα σε ό,τι συνιστά ευρωπαϊκή ε, μακροπρόθεσμη προστιθέμενη αξία. Άκουσα σήμερα το πρωί ότι υπάρχει συνένεση και ομοφωνία σε αυτό το τομέα. Θα πρέπει να δράσουμε όμως για να δράσουμε πραγματικά πρέπει να έχουμε όλες τις ίδιες προτεραιότητες και να δεχθούμε και περικοπές σε κάποιους τομείς. Στη γεωργία, ας πούμε, στη γεωργική πολιτική νομίζω επιβάλλεται μια τέτοια μείωση. Ε, ως ε, Σουηδικό Σοσιαλιστικό Κόμμα ε, φρονούμε ότι χρειάζεται όντως εξυγχρονισμός του προπολογισμού. Ετέθη το ερώτημα. Είναι όντως απαραίτητο ε, να ε, αφήνουμε τα κράτη-μέλη να μην επομίζονται τις ευθύνες τους. Υπάρχουν διάφορα επιχειρήματα εδώ. Βεβαίως να διευρυνθεί ο προπολογισμό να αυξηθεί, ε, γιατί υπάρχουν και χώρες που ε, ύφησαν τους προϋπολογισμούς τους τα τελευταία χρόνια πολύ περισσότερο από ό,τι αυξήθηκε ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Ε, ένας προϋπολογισμός θα πρέπει να είναι στραμμένος ε, στους συγκεκριμένους στόχους, αρμοδιότητες και εξουσίες που θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε. Σε όλες λοιπόν τις ανακοινώσεις και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της επικείμενης του Συμβουλίου αναφέρεται ότι χρειάζεται γενναία χρηματοδότηση και επένδυση στην απασχόληση. και κάθε πρόγραμμα σε ε, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο ε, περικόπτεται. Όλη, σε όλη την Ευρώπη βλέπουμε μια στάσιμη οικονομία. Η ενέργεια βρίσκεται σε καταστροφικά επίπεδα. Είναι επικίνδυνη η κατάσταση αυτή. Θέλουμε να αλλάξουμε αυτήν την καταστροφική πορεία. Αν ναι, υπάρχουν πέντε πράγματα που είναι σημαντικά. Καταρχήν, υπάρχει το θέμα του προϋπολογισμού, αλλά και η πολιτική της κρίσης θα πρέπει να διεξάγεται με πιο ισορροπημένο τρόπο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να υπάρχει κοινωνική διάσταση. Δεν μπορούμε να εφαρμόζουμε μόνο πολιτική λιτότητα. Θα πρέπει να έχουμε και πολιτική ανάπτυξη και πολιτική απασχόληση. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στην Ιρλανδία με τον κύριο Μπέρναρντ Ντάνκαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω εδώ και συμφωνώ με αυτή τη συγκέντρωση, τη συνάντηση των μελών του Εθνικού Κοινοβουλίου με τους συναδέλφους τους εδώ ώστε να κατανοήσουμε ένα τη θέση του άλλου. Ελπίζω ότι αυτό που θα προκύψει από αυτή τη συνάντηση θα είναι μια κατανόηση των θέσεων μας. Θα ήθελα να συγχαρώ τον συναδελφό μου, τον πρόεδρο Λίντσε για τη συμβολή του, πολύ χρήσιμη. Ελπίζουμε ότι θα την ακολουθήσουν οι Ευρωπαίοι συναδελφοί μας. Πολλά υπόθηκαν σήμερα το πρωί για την οικειοποίηση, το ownership και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να βρίσκεται στην καρδιά. Πάντα αναλαμβάνουμε ευθύνη όχι μόνο για τους δικούς μας προϋπολογισμούς αλλά και για τον προϋπολογισμό των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Και αυτό σημαίνει συντονισμένη οικονομική προσπάθεια. Σημαίνει επίσης ότι η κάθε χώρα έχει διαφορετικές ανάγκες. Άλλες πιο γεωργικές, άλλες πιο τεχνολογικές, άλλες ε, πιο βιομηχανικές. Ό,τι και αν είναι, πρέπει να είμαστε πάντα προσεκτικοί στην ε, Ιρλανδία. Εξαρτώμαστε ιδιαίτερα από τη γεωργία για να βγούμε από το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε. Και έτσι πράττουμε το 90% της παραγωγής μας πηγαίνει στις εξαγωγές σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει, να είχαμε επιτύχει όλα αυτά οικονομικά αν δεν είχαμε τη στήριξη της γεωργίας και πραγματικά επιμένω να διατηρηθεί. Αυτή η κακή οικονομική πολιτική μείωση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού ενώ ταυτόχρονα τα εθνικά κοινοβούλια αναγκάζονται να περικόψουν τους προϋπολογισμούς τους για λόγους που όλοι έχουμε συζητήσει. Δεν καταλαβαίνω γιατί μιλάμε συνέχεια για λιτότητα. Εγώ δεν την ονομάζω λιτότητα. Εγώ πιστεύω ότι μας ανάγκασαν απλά γιατί δεν είχαμε πόρους και έτσι χρειάστηκε να περικόψουμε τους προϋπολογισμούς μας. Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο για τους λαούς μας και υπάρχει δυσαρέσκεια, αλλά ξέρουμε ότι φέρνει αποτελέσματα. Αυτό όμως που χρειαζόμαστε είναι αναγνώριση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναγνωριστεί ότι αυτά που πράττουμε είναι σωστά. Χρειαζόμαστε υποστήριξη και χρειαζόμαστε και άλλες χώρες οι οποίες θα αναγνωρίσουν ότι προχωράμε μαζί στον ίδιο οδό. Ελείψη αυτού θα βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου μετά από 5 ή 10 χρόνια θα κάνουμε τις ίδιες ερωτήσεις. Θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα ίδια ζητήματα. Είναι πολύ σημαντικό κύριε Πρόεδρε να αναλάβουμε την ευθύνη μας αυτή τη στιγμή και να ενθαρρύνουμε τις χώρες που έχουν ήδη δείξει ότι είναι πολύ ισχυρέ σε συγκεκριμένους τομείς να κάνουν ό,τι μπορούν καλύτερα στον τομέα στον οποίο ειδικεύονται και με την υποστήριξη των συναδέλφων τους. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ συνάδελφε. Συγχαρητήρια στην Ιρλανδία για το παράδειγμα που δίνει Ο Πρωθυπουργό ήρθε τις προάλλες στο Κοινοβούλιο και μας ε, έδειξε τι συμβαίνει στη χώρα. Πολύ ενθαρρυντικό για όλες τις χώρες. Ε, τώρα ο εισηγητής ε, για την πολιετή δημοσιονομική συμφωνία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω κάποιες ανησυχίες προς τους συναδέλφους μας από τα Εθνικά Κοινοβούλια, διότι Πλησιάζει ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που μπορεί να λάβει αποφάσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό και τότε θα έχουμε προβλήματα εδώ στο Κοινοβούλιο, διότι θα πρέπει να πούμε ναι ή όχι σε αυτά που θα συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη. Και το θέμα με το Κοινοβούλιο είναι απλό. Αφενός ε, Προσπαθούμε να υποβάλουμε τα επιχειρήματά μας στο Συμβούλιο που μέχρι στιγμής δεν τα λάμανε υπόψη του. Να σας δώσω ένα παράδειγμα ε, για να καταλάβετε ότι το θέμα δεν είναι απλά ότι ζητάμε λεφτά. Πρέπει να έχετε κατά νου ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός ανέρχεται μάλλον φτάνει ε, το ένα πεντηκοστό των ε, εθνικών προϋπολογισμών. Πρόκειται για το 2% ε, των ευρωπαϊκών δημοσίων ταπανών. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά το μέγεθος του προϋπολογισμού. Η πρόταση που είχαμε τον ε, Σεπτέμβριο δεν, δεν επρόκειτο για πάγωμα. Ε, συνάδελφοι μας είπαν ότι παγώνουμε τον προϋπολογισμό. Όχι, ε, τον επαναφέρουμε ε, στο 2008 πριν την τελευταία διεύρυνση και ελπίζουμε ότι θα παραμείνει στα επίπεδα αυτά μέχρι το 2020. Δηλαδή, δεν παγώνουμε τον προϋπολογισμό τον επαναφέρουμε σε επίπεδα προηγούμενα του 2008 και του 2004 όπως ακούγεται και θέλουμε να διατηρηθεί μέχρι το 2020. Τα κράτη-μέλη λοιπόν αρνούνται να γίνει αυτό. Επίσης θέλουμε ε, περισσότερη ευελιξία. Κατά την έγκριση των εθνικών προπολογισμών θέλουμε με λιγότερα χρήματα να μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα. Αυτό όμω δεν μπορεί να γίνει αν δεν γίνουν αντίστοιχα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ο ευρωπαϊκό προπολογισμό ε, είναι πολύ πιο άκαμπτο από του ε, εθνικού προπολογισμού. Θα πρέπει να ληφθεί και αυτό υπόψη. Τρίτον, οι ίδιοι πόροι. Ο πρόεδρο Αλαμασούρ τον έφερε αυτό κατά την εισαγωγική του ε, παρέμβαση. Θέλουμε περισσότερη αυτονομία όσον αφορά του ίδιους πόρους, ώστε να μην βαρύνουν το, τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Ε, οι συμβολές λοιπόν προς, τους προς τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ε, ε, δεν θα επηρεάσουν τους εθνικούς προϋπολογισμούς, κάτι που θα είναι καλά νέα για όλους τους ε, υπουργούς οικονομικών. μιλάμε, δεν μιλάμε λοιπόν για περισσότερα χρήματα, μιλάμε για καλύτερη κατανομή. Και επίσης ε, όσον αφορά τις εξελίξεις ε, στην Ευρωζώνη, ιδιαίτερα την κατεύθυνση που έχει πάρει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, τώρα έχουμε νέες ε, ιδέες σχετικά με κάποιο νέο μέσο της Ευρωζώνης. Καλά όλα αυτά, αλλά εάν έχουμε πολλού διαφορετικού προπολογισμού, πάλι οι φορολογούμενοι θα πληρώνουν. Αυτό λοιπόν που θέλουμε είναι να έχουμε μια ενιαία εικόνα του ευρωπαϊκού προπολογισμού με τη δέσμευση όλοι οι φορολογούμενοι ε, να ε, ε, να καλύπτονται. Αυτό, αυτή είναι η δημοκρατική προσέγγιση, αυτό θέλει το Κοινοβούλιο. Αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο δεν δείχνει διατεθειμένο να απαντήσει στα αιτήματα αυτά και ανησυχώ ότι αν υιοθετηθεί με τέτοιο τρόπο η συμφωνία την επόμενη εβδομάδα δεν θα μπορέσουμε να την εγκρίνουμε εδώ στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε συνάδελφοι. Και τώρα από τη Μαύρη Θάλασσα περνάμε στην Βαλτική Πολωνία με τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Πολωνικής Βουλής, τον κύριο Γκαλαζεύσκη. Είναι... Όχι, δεν είναι εδώ. Με συγχωρείτε, δεν το πρόφερα σωστά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έρχομαι από τον νότο της Πολωνίας. Απέχει αρκετά από τη Βαλτική, η περιοχή μου. Παρόλο που έχουμε παράλια στην Βαλτική ως χώρα. Ο Επίτροπος Λεβαντόφσκι είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια πρωτόγνωρη θέση ο επόμενος προϋπολογισμός θα είναι μικρότερος από τον προηγούμενο, τους προηγούμενους. Επίσης, αυξάνονται οι υποχρεώσεις μας γιατί είναι πιο φιλόδοξοι οι στόχοι. Και οι δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει είναι πιο δύσκολο να επιτευχθούν. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ υπάρχουν κάποιες αντιφατικές τάσεις. Και θα ήταν καλό εάν μπορούσαμε να βρούμε έναν τρόπο να εξορθολογήσουμε τόσο τις υποχρεώσεις όσο και τους πόρους μας. Να κάνουμε δηλαδή περισσότερα με μειωμένο προπολογισμό. Αληθεύει ότι μας αναγκάζει ο μειωμένος προπολογισμός να βλέπουμε με τρόπο πιο επικριτικό και με περισσότερη κριτική σκέψη τις δαπάνες μας. Όμως ε, οι τάσεις που επικρατούν αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι που μας ικανοποιεί. Πώς λοιπόν να φέρουμε εις πέρα στις υποχρεώσεις μας. Θα συμφωνήσω εν μέρη με τον συνάδελφο από την ε, Ολλανδία. Όμως ο προπολογισμό θα εγκριθεί εντός των προσεχών εβδομάδων. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να προλάβουμε να τον προσαρμόσουμε, να τον εξυγχρονίσουμε. Ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020. Αυτό με βρίσκει απολύτω σύμφωνο ως επιλογή και για τα προηγούμενα θέματα που συζητήσαμε. Ο Επίτροπος Ρεν είπε ότι υπάρχουν σοβαρές αποκλήσεις μεταξύ των οικονομιών των κρατών μελών και γι' αυτό είναι τόσο σημαντική η πολιτική συνοχής για να έχουμε ισότιμους κανόνες παιχνιδιού σε ό,τι αφορά την κοινωνική ανάπτυξη και την απασχόληση στα κράτη-μέλη είναι απαραίτητο να αξιοποιηθεί, να αξιοποιηθεί η πολιτική συνοχή. Ευτυχώς έχει πολλούς υποστηρικτές που θα τις επιτρέψουν κατά πάσα πιθανότητα να επιβιώσει. Σε ό,τι αφορά την ερευνακή ανάπτυξη, είναι και αυτή μια πολύ σημαντική διάσταση. ως προς την ε, επιστημονική έρευνα, οι αποκλήσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες από ό,τι ως προς την οικονομική ανάπτυξη βάσει της μελέτης που έχουμε μπροστά μας. Ελπίζω ότι υπό το πρίσμα της Ευρώπης το 2020 αυτές οι αποκλήσεις θα περιοριστούν. και ότι κράτη-μέλη που δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμη ιδιαίτερως θα το βελτιώσουν αυτό. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ συναδελφέ και πάλι στην Ελλάδα ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, ο κ. Μπέζος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, αυτή η συνεργασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι μια συνεργασία απαραίτητη για να διασφαλιστεί η δημοκρατική νομιμότητα σε αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζουμε όμως ότι αυτή η συνεργασία στο μέλλον θα είναι πιο συστηματική και θα γίνεται με πιο ολοκληρωμένο τρόπο. Η Ελλάδα, όπως είναι γνωστό, βρίσκεται σε πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής και επομένως δεν είχε την υποχρέωση να καταρτήσει εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και πρόγραμμα σταθερότητας για το 2013. Παρά τα αυτά, κατέθεσε ένα ενημερωμένο εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, όπου παρουσιάζεται η μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνει η χώρα για μεταρρυθμίσεις και μάλιστα μια προσπάθεια η οποία γίνεται κάτω από συνθήκε ύφεση για πέμπτη συνεχή χρονιά σε κατάσταση ύφεση. Θα ήθελα να αφαιρθώ σε τρία πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Πρώτον, σε σχέση με την πολιτική συνοχή. Άποψή μα είναι ότι τα προτινόμενα στατιστικά στοιχεία για τη μεθοδολογία κατανομή των κονδυλίων αποκλίνουν σημαντικά από την υφιστάμενη σήμερα πραγματικότητα και σε καμιά περίπτωση δεν αποτυπώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις της ύφεσης. Επομένως, σε μια κρίσιμη περίοδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κρίσιμη για την ανάπτυξη και τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωση, η κατανομή των κονδυλίων της συνοχής βασίζεται, θα έλεγα, σε μια ξεπερασμένη εικόνα τη οικονομία των κρατών μελών και των περιφερειών του. Εμεί θεωρούμε ότι το μέγεθο τη μείωση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντο σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη άνοδο των ποσοστών τη ανεργία εντό των κρατών μελών θα πρέπει να ληφθούν οπωσδήποτε υπόψη όταν θα γίνουν οι τελικέ ρυθμίσει στι μεθόδου κατανομή των πόρων τη συνοχή. Η δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει με τον τομέα τη έρευνα. Ο τομέα τη έρευνα και τη καινοτομία είναι όντω πολύ σημαντικό για τη βελτίωση τη ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών, όχι μόνο σε επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε διεθνέ επίπεδο. Παρόλα αυτά όμω, η μείωση των αναγκαίων πόρων, και η υποβάθμιση τη πολιτική συνοχή θα έχει σαν αποτέλεσμα κράτη-μέλη και περιφέρειες οι οποίε βρίσκονται σε κατάσταση ύφεση να μην μπορούν να προχωρήσουν σε αναπτυξιακέ επενδύσει. Πρέπει επομένω αυτό να το λάβουμε υπόψη μα, να λάβουμε δηλαδή υπόψη μα ότι η ενίσχυση τη εξωτερική ανταγωνιστικότητα τη Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρί την εμβάθυνση τη εσωτερική τη συνοχής. Και η τρίτη παρατήρηση έχει να κάνει με το σκέλο των εσόδων. Ε, πιστεύουμε ότι η κύρια πρόκληση την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στη δημιουργία ενός μείγματο ιδίων πόρων για την επαρκή χρηματοδότηση των κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών, όπως ο φόρος για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές ή ο ευρωπαϊκός φόρος προστιθέμενης αξίας και από την άλλη μεριά η παράλληλη μείωση της επιβάρησης των προπολογισμών των κρατών μελών. Αυτή όμως αυτό το σύστημα εφαρμογή των ιδίων πόρων θα πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αποτελεσματικό στη λειτουργία του και να μην δημιουργεί επιπρόσθετο κόστο διοικητική διαχείριση. Σα ευχαριστώ πολύ. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Ήταν ιδιαίτερο ενδιαφέρουσα η εισήγησή σα. Επιστρέφουμε στην Ιρλανδία και δίνω το λόγο στον βουλευτή, κύριο, στον γερουσιαστή κύριο Λάιντεν. Είναι μέσα στην αίθουσα. Όχι. Δεν θα πάρει το λόγο. Επιστρέφουμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο κύριος Γκαρίγκα. Ελσενιόρ Γκαρίγκα. Eh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζω ότι οι εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων που παρευρίσκονται σήμερα εδώ έχουν έντονο φιλοευρωπαϊκό χαρακτήρα και στα κοινοβούλια τους είναι καμιά φορά πιο δύσκολο να υπερασπιστεί κανείς τη φιλοευρωπαϊκή του στάση από ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εδώ όμως που φτάσαμε και συζητούμε θα πρέπει να μας απασχολήσει το εξής. Εσείς πιστεύετε και τα εθνικά σας κοινοβούλια ότι ο κοινοτικό προϋπολογισμός είναι έκφραση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας ή όχι. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτή η πεποίθηση στα εθνικά κοινοβούλια και θεωρείται ο κοινοτικός προϋπολογισμός ως ένας επιπρόσθετος, 29ος βάζω και την Κροατία μέσα, ε, εκτός των εθνικών, τότε θα μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι θα υποστηρίζετε τις κυβερνήσεις σας να υπογράψει για μια ευτετία ένα προϋπολογισμό με 22 δισεκατομμύρια χαμηλότερο από τον τρέχοντα. Σε περίπτωση όμως που εσείς πιστεύετε κάτι διαφορετικό για τον κοινοτικό προϋπολογισμό, ότι είναι δηλαδή σημαντικό ε, να υπερασπιστείτε και στα εθνικά σας κοινοβούλια κάποιες άλλες ε, προτάσεις ότι έχει κάποια περιορισμένη αντικυκλική ε, λειτουργία ή σε βραχυπρόθεσμη ε, δημοσιονομική προσαρμογή ε, μόνο ο κοινοτικό προϋπολογισμός μπορεί να φέρει επενδύσεις μέσω και μακροπρόθεσμες. Αν λοιπόν αυτό πιστεύετε, αν πιστεύετε ότι ορίζον 2020 είναι μια ευρωπαϊκή ατζέντα ανάπτυξης που αξίζει σωστή χρηματοδότηση, εάν πιστεύετε ότι οι υποχρεώσεις που υπέγραψε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ενέκρινε το Εθνικό Κοινοβούλιο, κύρωσαν τα Εθνικά Κοινοβούλια, αξίζουν τον κόπο να υλοποιηθούν. Αν συμβαίνουν όλα αυτά, τότε θα πρέπει να προβληματιστούμε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε ως ευρωβουλευτές για να πείσετε εσείς τις κυβερνήσεις σας και τη Βουλή ε, του ο καθένας όπου γίνεται ότι δεν θα πρέπει τα πάντα να τα βλέπουμε ε, από τη σκοπιά των εθνικών συνεισφορών σε ένα κοινοτικό προϋπολογισμό αλλά να έχουμε υπόψη μας και την επιτυχία των κοινών πολιτικών. Είτε είναι αυτές πολιτικές καινοτομία, γεωργίας, συνοχής, εξωτερικής δράσης, κάθε ένα από τους τομείς που αφορούν τον κοινοτικό ε, προϋπολογισμό και ε, που επιβάλλεται να εγκριθεί για την επόμενη επταετία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κάνει αυτή την προσπάθεια και μπορείτε κι εσείς κάλλιστα να διαβιβάσετε τη γνώμη του Κοινοβουλίου μας στην εκάστοτε Βουλή του καθένα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Θα δώσω τώρα το λόγο εξ ονόμα της Συμβουλής των Λόρδων στη Βαρόνη Οκάφιν. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. έχει αναφερθεί επανειλημμένα η ανάγκη για την έρευνα και ανάπτυξη για να δώσει ορμή στην ανάπτυξη. Αλλά ο προϋπολογισμός του ορίζον 2020 ε, και του ε, πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου ε, οι σχετικέ διαπραγματεύσει μάλλον ήταν πολύ μακρέ, διέκυσαν πολύ, κάτι το οποίο μάλλον έχει οξυνθεί από την οικονομική κρίση. Ε, έχοντας αυτό κατά νου, ποιες προκλήσεις πιστεύετε ότι συνδέονται με την ε, χρησιμοποίηση του προϋπολογισμού, με τη χρήση του προϋπολογισμού για την ε, έρευνα και ανάπτυξη, διότι είναι πολύ δύσκολο για τα κράτη-μέλη να υπολογίσουν την απόδοση των σχετικών επενδύσεων. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να γνωρίζουμε τι μηχανισμούς χρησιμοποιεί η Κομισιόν ε, για να υπολογίσει την σχέση κόστους-όφελους ε, αντί για να χρησιμοποιούμε το κανονικό μοντέλο που χρησιμοποιούν επιχειρήσεις. Και μια δεύτερη ερώτηση που δεν συνδέεται άμεσα με αυτήν, αλλά ε, όπως ανέφερε μέλος των Γερμανών Πρασίνων για τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, θα ήθελα να ρωτήσω εάν η Κομισιόν έχει ασχοληθεί περαιτέρω με τις επιπτώσεις ε, στον προϋπολογισμό, με τη μελέτη επιπτώσεων που έχει γίνει για τον προϋπολογισμό. Σε πρόσφατη μελέτη επιπτώσεων η Κομισιόν κατέληξε ότι η πρότασή της δεν βοηθάει ιδιαίτερα στην ε, ε, δημιουργία ίδιων πόρων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Βαρόνη. Δίνω τον λόγο στον πρόεδρο Τζανκαλο Τζοτζέτη της Επιτροπής Προεπολογισμού του Ιταλικού Κοινοβουλίου. Κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι εκτίμησα ιδιαίτερα σήμερα το πρωί την ομιλία του κυρίου Μαρινή. Ήταν πολύ ειλικρινής. Το ίδιο θα ήθελα να είμαι και εγώ. Δεν συμμετέχω για πρώτη φορά σε συναντήσεις αυτού του είδους και Πρέπει να πω ότι δυστυχώς η προσπάθεια για να προσδοθεί δημοκρατική νομιμότητα στις αποφάσεις και τον προπολογισμό. Ειδικότερα θεωρώ ότι ειλικρινά είναι δύσκολο να επιτύχει. Δεδομένης της πραγματικής ε, ανάδυσης προβλημάτων οικονομικών και απασχόλησης, τα πράγματα που ξέρω σήμερα το πρωί ε, πρώτα από τους δύο επίτροπους και με τα, θέματα για τον κοινοτικό προϋπολογισμό μου φαίνονται όλα τα επιχειρήματα πολύ αδύναμα, ανεπαρκή. Έτσι η νομιμοποίηση αυτή που φτάνει μέχρι εμάς τους εθνικούς βουλευτές και στο λαό δεν φαίνεται να έχει σωστή υπόσταση. Εγώ μιλώ ω πρόεδρος της Επιτροπής Προπολογισμού, αλλά ξέρετε όλοι ότι στην Ιταλία τα πράγματα θα αλλάξουν σύντομα. Θα μπορούσα να μιλήσω κι εγώ λοιπόν και ως πολίτη Χθε συμμετείχα σε μια συνέλευση μικρών και μεσαίων επιχειρηματιών. Αύριο ίσως θα συμμετέχω σε κάποια άλλη. Μπορώ να σα πω ότι το κοινό αίσθημα, τα κοινά αισθήματα διαφέρουν όσον αφορά τις δράσεις στην Ιταλία, στην Ευρώπη δεν υπάρχει έτσι κοινή αίσθηση νομιμότητας. Υπάρχει ένα πρόβλημα νομιμότητας ε, ενώπιον των Εθνικών Κοινοβουλίων εκ μέρους του λαού. Για να σας δώσω την αίσθηση που αποκόμισα εγώ χθε και που θα αποκομίσω και αύριο, μου είπαν για ποιο λόγο το δημοσιονομικό σύμφωνο μας ε, οδηγεί σε φορολόγηση μεγαλύτερη της εργασίας, ενώ στην Ευρώπη δυσκολεύονται να μιλήσουν για φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που θα μπορούσε να χρηματοδοτεί τον ε, ε, κοινωτικό προπολογισμό. Γιατί στέλνουμε χρήματα στην Ευρώπη που μας έρχονται πίσω μέσω των διαφορών ταμείων, όπως είπε ο κ. Λεβαντόφσκι. Εμείς οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες δυσκολευόμαστε να έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα κονδύλια λόγω της γραφειοκρατίας δεν είναι εύκολη η συμμετοχή μας ε, χωρίς ιδιαίτερη βοήθεια. Τρίτη παρατήρηση. Μιλάμε για τα μεγάλα ζητήματα. Δυσκολευόμαστε ακόμη και να επικυρώσουμε τον ετήσιο προπολογισμό της Ένωσης. Για να ολοκληρώσω πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αποφασίσει για τα μεγάλα ζητήματα, τα οικονομικά, αλλά δυσκολεύεται να κάνει επεμβάσει στην πραγματική οικονομία. Για την η οικονομία μπορούμε να αποφασίζουμε, για την απασχόληση θα πρέπει να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετικά σημαντική η παρατηρήση σας, κυρία Άλντα Σούζα, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Πορτογαλίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να χαιρετήσω όλους τους ε, βουλευτές και ευρωβουλευτέ που βρίσκονται σήμερα σε αυτή τη διάσκεψη. Τέθηκαν πολλά ζητήματα, πρώτα απ' όλα από τον κύριο Λεβαντόφσκι, αλλά και από συναδέλφους μου και του Ευρωκοινοβουλίου. Για τον ε, ευρωπαϊκό προπολογισμό και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν βρισκόμαστε σε κατάσταση παγώματος, αλλά σε απειλή σοβαρής μείωσης, βίαιης θα έλεγα. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και ο ετήσιος και ο πολιετής είναι ισχνός, δεν είναι αρκετά φιλόδοξος, είναι θα έλεγα μινιμαλιστικός και πολλές φορές κάτω από τα κατόφλια και τα όρια που προβλέπουν οι ίδιες οι συνθήκες ορίζονται και κάποιες βασικές τιμές στις συνθήκες. Έτσι, αυτός ο προπολογισμό δεν διασφαλίζει την αναδιανεμητική λειτουργία και την ε, απόδειξη της αλληλεγγύης. Εμείς θα ήμασταν υπέρ της αύξησης του ευρωπαϊκού προπολογισμού και βεβαίως της αύξησής του και στο πολιετές επίπεδο. Εδώ υπάρχουν ευθύνες κοινέ για τους ευρωβουλευτές και για τους εθνικούς βουλευτές, διότι στο κάτω-κάτω της γραφής το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο με την παρουσία των κυβερνήσεων ε, έχουν επιδοθεί σε ένα μπραντεφέρ, σε ένα διαγωνισμό δύναμης. Εδώ θα έπρεπε και τα εθνικά κοινοβούλια να έχουν ε, λόγο στο όλο θέμα και μάλιστα να ακούγεται η φωνή τους γιατί είναι σοβαρά πολιτικά ζητήματα αυτά που μας απασχολούν. Θέλω να κάνω και άλλες δύο-τρεις παρατηρήσεις. Πρώτον, δεν νομίζω ότι είναι σωστό να λέμε ότι η οικονομική κρίση επέβαλε την λιτότητα. Η λιτότητα υπήρξε πολιτική επιλογή και μάλιστα επιλογή των ίδιων των ε, χωρών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα προγράμματα προσαρμογής στα οποία έχουν υποβληθεί κάποιες χώρες καταστρέφουν την απασχόληση και την ε, ανάπτυξη και προκαλούν ε, κοινωνική καταστροφή. Σε σχέση με τον προπολογισμό, η δική μας προοπτική είναι ότι ο φόρο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών είναι ζωτική σημασία. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν υπάρχουν ήδη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε είναι θεμελιώδη σημασία για τι μακροπρόθεσμε επενδύσει που σχεδιάζουμε, αλλά είναι και θέμα κοινωνική δικαιοσύνη. Γιατί είναι αναγκαίο να αυξήσουμε και το οικονομικό μα κεφάλαιο. Και έπειτα ω προ την έρευνα και ανάπτυξη, εδώ έχει γίνει λόγος για την κινητικότητα. Προφανώς η κινητικότητα των Ευρωπαίων πολιτών είναι άκρο σημαντική εφόσον είναι εθελοντική, δηλαδή προσωπική επιλογή, αλλά εφόσον είναι καταναγκαστική είναι κάτι τελείω διαφορετικό. Εδώ θέλουμε θέσει εργασία, επιστημονική έδρε έρευνα, οι οποίε δυστυχώ ακόμα είναι επισφαλεί για όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού βίου. Δεν παρέχουν καμία σταθερότητα στην ζωή των επιστημόνων. Να δημιουργήσουμε θέσει εργασία, λοιπόν επιστημονικέ, σταθερέ και μακροπρόθεσμε πρόεδρο. ευχαριστούμε συνάδελφε. Κοιτάξτε, συνάδελφοι, έχουμε πίεση χρόνου. Ακόμη πέντε αγορτέ έχουν ζητήσει το λόγο. Δεν μπορώ να του τον δώσω, λυπάμαι. Λοιπόν, Κύριε Γερουσιαστά, λάβατε το λόγο μια φορά το πρωί. Και θα μπορέσετε και το απόγευμα. Αλλά Με συγχωρείτε κύριε Γερουσιαστά, δεν μπορώ να σας το επιτρέψω αυτό. Ε, μιλήσατε το πρωί. Σημειώσαμε και τις παρατηρήσεις σας, οι οποίες ήταν εύστοχες, αλλά τουλάχιστον άλλοι έξι συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο, δεν πήραν το λόγο το πρωί. Δυστυχώς, οι διερμηνείς θα πρέπει να φύγουν στη μία η ώρα. Υπάρχουν κάποιες ε, κάποιοι περιορισμοί και πρέπει να γίνουν περικοπές χρόνου, όπως γίνεται με τον προπολογισμό. Είναι κάποιες ε, περικοπές από αυτές, είναι λίγο αντιφατικές. Θα σας δώσω λίγα λεπτά παραπάνω και ευχαριστώ τους διερμηνείς που θα μείνουν μαζί μας για λίγο ακόμη, μετά τη μία. Και θα παρακαλέσω και τον Επίτροπο να απαντήσει εντάχει στις βασικές παρατηρήσεις που έγιναν και μετά η κυρία Τρότμαν θα κλείσει την πρωινή μας συζήτηση. Κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ. Είναι δύνατο να απαντήσω σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά θα προσπαθήσω. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι για να ε, έχει ε, νομιμότητα αυτή τη στιγμή η Ευρώπη θα πρέπει να ε, λύσει τα προβλήματα των ανθρώπων. Και είμαι Βεβαίως ότι υπό τους παρόντες περιορισμούς ε, οι στους εθνικούς προϋπολογισμούς ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός ε, μπορεί να βοηθήσει, όχι όμως με οποιοδήποτε τίμημα, γι' αυτό θα πρέπει να υπερασπιστούμε το επίπεδο των πληρωμών και θέλω να υπερασπιστώ την ε, την σύγκριση που γίνεται ανάμεσα στους εθνικούς προϋπολογισμούς και τον ευρωπαϊκό, ε, κάτι που αμφισβήτησε ε, ο κ. Πενχάρτσον από τη Σουηδία, διότι ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την διεύρυνση μέχρι το 2010 είχαμε περιορισμού στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, αυξήθηκε λιγότερο από ό,τι οι εθνικοί προϋπολογισμοί. Παρότι το ε, χρονικό διάστημα αυτό ε, έγινε χωρίς αρμοδιότητων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, η Σουηδία και η Γερμανία είναι οι, μόνοι, είναι οι μόνες εξαιρέσεις. θα, ήθελα όμως με τη σύγκριση αυτή να σας δείξω ποιοι είναι οι περιορισμοί της Ευρώπης. εξυγχρονισμός, ναι. Αυτό περιλαμβανόταν στην αρχική μας πρόταση του 2011, αλλά όπως είπαν ε, αρκετοί ομιλητές, η ε, Χέλγα Τρούιπελ, ο κύριος Κάλφιν και άλλοι, εάν γίνουν περικοπές, αυτές ε, οφείλονται περισσότερο στη λογική των διαπραγματεύσεων. Υπάρχουν χώρες που ακόμα ζητάνε πιο βαθιές περικοπές. Μας ενδιαφέρει ο εξυγχρονισμός, η προστιθέμενη αξία, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε τη λογική, ε, διότι δεν μπορούμε ταυτόχρονα να ζητάμε περικοπές ε, στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ωστόσο, Ωστόσο, όλοι ήταν υπέρ ε, του να ε, ενισχυθεί η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ε, είναι δυνατόν με λίγα χρήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να διατηρούμε δύο εκατομμύρια ανθρώπους ε, στα, στους καταβλισμούς προσφύγων ε, στη Συρία. 1,5 εκατομμύριο ανθρώπων ε, στο Ιράκ. Ε, πάλι έχουμε μικρό, μικρό ποσό χρημάτων ε, που έχει συγκεντρωθεί από διάφορα κράτη-μέλη και έτσι πετυχαίνουμε σημαντικό αποτέλεσμα. Δεν περιμένουμε κάποια επανάσταση στην πλευρά των εσόδων. θέλουμε μάλλον ενισχυμένη συνεργασία. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί απέναντι σε ένα πιο λαμπρό μέλλον ε, με τον ε, ε, φόρο επί των οικονομικών συναλλαγών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε το το Νόμπελ Ειρήνης ε, για το παρελθόν της ε, και νομίζω ότι της αξίζει. Άλλωστε είχαμε οικονομική ειρήνη τα τελευταία 7 χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, η κυρία Τροτμάν, εισηγήτρια στην Επιτροπή Προπολογισμών. Ευχαριστώ πρόεδρε, με λίγα λόγια και πολύ σύντομα. Πρώτον, νομίζω πρέπει να καταγράψουμε ότι συλλογικά οι Ευρωβουλευτέ και οι Εθνικοί Βουλευτέ επέμειναν στο γεγονό ότι ο προπολογισμό μα είναι ένα προπολογισμό των 28. Όχι ένα προπολογισμό που πρέπει οι μεν να αποφασίζουν και οι δεν να εφαρμόζουν. Δεν μπορεί έτσι ο προπολογισμό μα να αναλάβει το ρόλο του μοχλού τη μόχλευση τη οικονομική ανάπτυξη. Έπειτα για την ετήσια επισκόπηση τη ανάπτυξη θα πρέπει, ε, είναι επιτακτική ανάγκη να επιτρέψει αυτή η επισκόπηση να δώσει τον πλήρη ρόλο του στον ευρωπαϊκό προπολογισμό με καταλητικό ρόλο για την χρηματοδότηση και με συμπληρωματικό ρόλο για την ίδια. Εδώ η επισκόπηση αυτή μπορεί να δώσει μια άλλη διάσταση στον ευρωπαϊκό προπολογισμό με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη και την ε, Απασχόληση. Μια άλλη παρατηρήση που καταγράφω από την όλη συζήτηση είναι οι συστάσει αναχώρα και οι συνεισφορέ των κρατών μελών. Είπατε, Πρόεδρε, ξεκινώντα την ε, μεσημεριανή μα συζήτηση και σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό, ότι σήμερα υπάρχει ανισότητα ανισότητα στον τρόπο που τα κράτη-μέλη συνεισφέρουν στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Αυτό το σημείο πρέπει να εξεταστεί. Ιδάλλως, διαρκώς θα υπάρχει τάση μείωσης των συνεισφορών των κρατών μελών στον προπολογισμό της Ένωσης. Αυτό μας οδηγεί σε αδιέξοδο. Αδιέξοδο δημοσιονομικό του προπολογισμού και ίσως να μας οδηγήσει και σε αδιέξοδο σε επίπεδο δημοσιονομικών προοπτικών. Η δική μου η πρόταση ήταν από από τον υπολογισμό των εθνικών ελλημάτων να αφαιρέσουμε τις συνεισφορές τους για την έρευνα και ανάπτυξη. Και τα κράτη-μέλη ε, καταψήφισαν σε μια πρώτη φάση, όμως ελπίζουμε να προχωρήσουμε σε αυτόν τον δρόμο. Διότι ο ευρωπαϊκός προπολογισμός είναι προπολογισμός επενδύσεων, οπότε εφόσον θέλουμε να ανακάμψει η ανάπτυξη με επενδύσεις, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε ουσιαστικά ποινέ σε κράτη-μέλη που είναι δικαιούχοι υπό το ίδιο πρίσμα και ω προς τον εκδημοκρατισμό. Η δημοκρατική νομιμοποίηση πρέπει να επιτρέψει στα κράτη-μέλη, στα Εθνικά Κοινοβούλια και στο Ευρωκοινοβούλιο να συνεργάζονται υπό την προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και εδώ να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω λέγοντας ότι καλό θα είναι να πετύσουμε από τα κράτη-μέλη και κάποια συνοχή. Νομίζω η συνοχή είναι και το κλειδί για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Όταν τα κράτη-μέλη, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν εμείς οι ίδιοι ευρωβουλευτές διατυπώνουμε φιλόδοξους στόχους και βλέπουμε ότι δεν έχουμε τα απαραίτητα μέσα, ουσιαστικά χάνουμε την αξιοπιστία μας και την ε, δημοκρατική μας νομιμοποίηση. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο η Επιτροπή μας ήταν, έδειξε ιδιαίτερη πυγμή στο σημείο αυτό, στο ότι τα κρατη να πληρώσουν ε, τους λογαριασμούς τους. Πώς να πληρώσουν λογαριασμούς όμως, εάν δεν έχουμε προπολογισμούς που να είναι κατάλληλοι και για τις πολιτικές μας. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε πρόβλημα χρηματοδότησης. Δεν μπορούμε λοιπόν ε, να απαιτούμε από τα κρατη να πληρώνουν τα χρέη τους, τα δημόσια χρέη, και αυτά στο επίπεδο και στην κλίμακα του προπολογισμού. Αυτές ήταν οι καταληκτικές μου παρατηρήσεις, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφε. Θα ήθελα για να ολοκληρώσουμε τι εργασίε μα, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, να σα ευχαριστήσω όλου για τη συμμετοχή σα. 16 ομιλητέ, είχαμε κατά τη διάρκεια αυτή τη συνεδρίαση, ε, αυτού του εργαστηρίου, μετά από την λίγο δυσάρεστη παρατηρήση του συναδέλφου από τη Γαλλική Γερουσία, θα ήθελα να σα πω ότι κανένα μέλο σήμερα το πρωί δεν μπόρεσε να μιλήσει δύο φορέ αφενός και αφετέρου υπάρχει τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος κάθε εθνοσυνέλευσης που ζήτησε το λόγο και που τον έλαβε. Από όσο γνωρίζω, εκτός αν κάποιος έχει αντίθετη άποψη. Και στην περίπτωση της Γαλλίας η Εθνοσυνέλευση, η Γερουσία και τα δύο σώματα της Γαλλίας είχαν κάποιον ομιλητή ο οποίος πήρε το λόγο σήμερα το πρωί. Φυσικά υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι ήθελαν να μιλήσουν σήμερα το πρωί, οι οποίοι δεν κατάφεραν, οι διερμηνεί χρειάζεται να φύγουν, δυστυχώ δεν μπορούν να μιλήσουν αυτή τη στιγμή, θα έχουν προτεραιότητα εφόσον επιθυμούν να μιλήσουν σήμερα το απόγευμα. Το επισημαίνω αυτό στου ε, συνάδελφου μου που θα προεδρεύσουν τη συνεδρία σήμερα το απόγευμα. τέλο, για να ολοκληρώσουμε με μια ευχαριστηνότητα, με μια καλή είδηση. Φυσικά Όλοι σας είστε προσκεκλημένοι τώρα κατά το μεσημεριανό διάλειμμα στο γεύμα που θα λάβει χώρα η συγγένεια των Εθνικών μας Κοινοβουλίων και των προϋπολογισμών μας. Καλή σας όρεξη. Διακόπτη συνεδρίαση μέχρι σήμερα το απόγευμα.